Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μας ε, δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα ε, των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΠΑ ΕΕ, για την δεύτερη συμφωνία για τις και κυκλοφορίες. Το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη συμφωνία σε δεύτερο στάδιο, μια συμφωνία την οποία υποστήριξε στεναρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαδραμάτισε και πολύ επικοδομητικό ρόλο στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευγνώμων. Να σταθώ στα βασικά στοιχεία αυτής της ε, συμφωνίας σε δεύτερο στάδιο. Η συμφωνία αυτή προσθέτει στοιχεία στην ε, συμφωνία σε πρώτο στάδιο, από τις, ε, που έγινε στις 30 Μαρτίου του 2008 για δημιουργώντας νέες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά καθώς επίσης και ενισχύοντας περαιτέρω την συνεργασία για ρυθμιστικά θέματα όπως για παράδειγμα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής προστασίας, ανταγωνισμού και ασφάλειας. Ως προς το περιβάλλον, το σχέδιο συμφωνίας σε δεύτερο ε, στάδιο καθορίζει ένα πολύ στενερό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις ε, που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω κοινών προγραμμάτων, εφαρμογής πρακτικών λύσεων, παραδείγματος χάρη ε, καθαρές τεχνολογίες ε, εναέριων τεχνολογιών, όπως και συνεργασία πολιτικών υπηρεσιών αεροπορίας. Επίσης, ε, αναγνωρίζεται η σημασία του να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και ο καθένας ε, να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα μέτρα του ε, για την αγορά, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφαληθεί από την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της ασφάλειας. Η συμφωνία προσπαθεί να μειώσει το... Ε, άχθος που υπάρχουν στα αεροδρόμια για θέματα ασφαλείας και ε, κάνοντας και κατάλληλες διαβουλεύσεις για τις μελλοντικές απαιτήσεις. Σε θέματα ανταγωνισμού ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς επίσης και η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα των αποφάσεων πλαίσιο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και για πρώτη φορά σε μια τέτοια συμφωνία και κυκλοφορίας αναγνωρίζεται η ανάγκη να εξισορροπηθούν οι ε, δυνατότητες που προσφέρονται στην αγορά με τις κοινωνικές ε, προκλήσεις κατά τρόπον ώστε να μην ε, υπονομεύονται τα εργατισιακά δικαιώματα. Σε εμπορικό επίπεδο η Ευρώπη έχει αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα ε, έχει άμεση πρόσβαση στο Fly America Program με την εξαίρεση των θεμάτων της άμυνας. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι τώρα χρηματοδοτούσαν αέριες μεταφορές μόνο ε, αμερικανικών αεροπορικών εταιριών. Και υπάρχουν και δεσμεύσεις για να προχωρήσουμε περαιτέρω ως τμήμα της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ έχουν δεσμευθεί ώστε να άρουν τους υπόλοιπους φραγμούς που υπάρχουν για το εμπόριο, καθώς όπως για παράδειγμα αυτούς που ε, δεν επιτρέπουν τη σωστή πρόσβαση σε κεφάλαια. Η πρόοδος θα εξετάζεται ετησίως και θα προχωρούμε από κοινού μέσω της κοινή επιτροπής. Θα υπάρχει και μία αναθεώρηση σε υψηλό επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη πρόοδος, έχουμε ε, καθορίσει και συγκεκριμένους στόχους για να προχωρήσει ο τομέας αυτός και οι δύο πλευρές ε, θέλουν να προχωρήσει ο τομέας αυτός ε, και να υπάρχουν και τα δικαιώματα επιβατών ε, και η κυκλοφορία σε τρίτες χώρες. Συνοπτικά, η Συμφωνία προχωρεί τα θέματα της συνεργασίας σε ένα μεγάλο φάσμα ρυθμιστικών θεμάτων, όπως θέματα ασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών και περιβάλλον έχει άμεσες και μελλοντικές επιπλέον ε, δυνατότητες εμπορίου και ε, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για μεταρρυθμίσεις καθώς επίσης ενισχύει την υπάρχουσα συμφωνία σε πρώτο στάδιο η οποία θα είναι ενισχύ εάν δεν ε, θα χαθεί συγγνώμη αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία σε δεύτερο στάδιο. Έχουν γίνει εκτιμήσεις ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μέχρι και 12 δις ευρώ σε οικονομικά ωφέλη και καθώς επίσης και 20.000 νέες θέσεις εργασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, σε αυτό το νέο οικονομικό κλίμα. Ελπίζω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία. Σα Σας κατευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο για τους επόμενους στους εκπροσώπους πρώτα των πολιτικών αμάδων. Πρώτα ο κύριος Ματθαίος Γκρός, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Συμφωνία Εναερίων Μεταφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ασφαλώς σημαντική. Για τον λόγο αυτό νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήγαγε ζωηρότατες συζητήσεις. 60% των συνολικών αερίων μεταφορών παγκοσμίω είναι η κίνηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένης Ευρώπης. Ελπίζουμε και οι δύο πλευρές να αντιληφθούν την ανάγκη γνήσιας διμερού συμφωνίας και ελπίζω και στο μέλλον να τους ενθαρρύνεται για μια συνεχή βελτίωση με κάθε σεβασμό για την εργασία που επιτελέσατε και βεβαίως και με όλο τον θαυμασμό που διαθέτω για την αισιοδοξία των διαπραγματευτών σας, θεωρεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι μένουν ακόμα ορισμένα πράγματα που πρέπει να διαπραγματευτείτε και ότι ίσως δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο ικανοποιημένοι με το παρόν αποτέλεσμα. Είχαμε ορισμένα εκκρεμή θέματα, αφενός η κεφαλαιακή συμμετοχή ελπίζαμε να επιτευχθούν κάποιες πρόοδοι. Για να είμαστε ειλικρινείς πρόοδοι δεν υπάρχουν σχεδόν. Το μόνο που έχουν πει είναι ότι θα συζητήσουν. Δεύτερο, οι υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου που είχαμε και εκεί πει ότι πρέπει να υπάρξουν πρόοδοι προς το κοινό συμφέρον, προς το αμοιβαίο συμφέρον. Ούτε εκεί είδαμε τέτοιες πρόοδους. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά δεν τολμούμε καν να μιλήσουμε για καμποτάζ φαίνεται να μην συζητείται κάτι τέτοιο από πλευρά Πολιτειών. Εμείς πρέπει να δούμε το στοιχείο της αμοιβαιότητα που δεν έχει επιτευχθεί απολύτω. Ό,τι δηλαδή προσφέρουμε στους άλλους πρέπει να το απολαμβάνουμε και εμείς. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν υποτιμούμε όπως το, η κοινωνική διάσταση κατά τα λοιπά όμως δεν επιτεύθηκαν μεγάλες πρόοδοι. Βέβαια αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η θέληση για να επιτευχθούν πρόοδοι στο μέλλον. Θα σημειώσω τρία σημεία σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Πρώτο, χρειάζεται μια νομική βάση για τέτοιε συμφωνίε και κυρίω για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Νομίζω ότι εκεί χρειαζόμαστε νομοθετική ρύθμιση και τήρηση κυρίω τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και εν πάση περιπτώσει να μην τεθεί το Κοινοβούλιο ενώπιον τετελεσμένων γεγονότων. Δεύτερον, να τονιστεί ο αμοιβαίος χαρακτήρας των συμφωνιών αυτών. Όχι μόνο μερίς, αλλά αμοιβαίος, διμερής χαρακτήρας. Τρίτο, να καθοριστεί η ημερομηνία για την επανέναρξη νέων διαπραγματεύσεων. Είπατε ότι κάτι θα γίνει μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2010. Αλλά ελπίζω ότι από κάθε άποψη και οικονομική και κοινωνική και περιβαλλοντική θα καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία στο όχι πάρα πολύ απομακρυσμένο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ελχαντράουι, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το 2007 καταλήξαμε σε συμφωνία για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων με, για τις αεροπορικές μεταφορές και η έννοια του ευρωπαϊκού μεταφορέα έγινε τότε δεκτή. Οπουδήποτε δηλαδή υπήρχε μια εταιρεία που είχε το δικαίωμα να πετάξει από την Ευρώπη μπορούσε να πάει οπουδήποτε στις ΗΠΑ. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, Μία μεικτή επιτροπή είχε συσταθεί για να υπάρχουν τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν τις θέσεις τους και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και τελικά μία πραγματική κοινή αερομετα... Ε, αγορά αερομεταφορών από τις δύο πλευρές αλλά οι Αμερικανοί είχαν περισσότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από ό,τι το αντίθετο. Και φυσικά υπήρχε πολύ μικρότερη συμμετοχή στα κεφάλαια των Ευρωπαίων. Και γενικότερα είχαμε συμφωνήσει στα τέλη του έτους να κάνουμε μια ενημέρωση, να ζητήσουμε περισσότερες παραχωρήσεις από τους Αμερικανούς Έχουμε μπροστά μας ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραμένουν οι ανισότητες και οι ελλείψεις και δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος για την καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς και στον έλεγχο των κεφαλαίων και την ιδιοκτησία των εταιριών. Παρά τα λίγα θετικά στοιχεία λοιπόν που ανέφερε και προηγούμενο συνάδελφος, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας εκτός εάν γίνει περισσότερη πρόοδο στο μέλλον και μπορέσει να δοθεί η εγγύηση ότι θα υπάρξει περισσότερη πρόοδο ως προς τα δικαιώματα των επιβατών και την πρόσβαση στις αγορές των αερομεταφορών. Αυτό θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση για να κάνουμε και εμείς περαιτέρω παραχωρήσεις στους Αμερικανούς. Ελπίζω δε η Κομισιόν να μα στηρίσει πλήρω ενήμερου για, ε, ε, για την πρόοδο των για να ξέρουμε και εμεί τι ακριβώ συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μάισνερ εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, παρουσιάσατε την συμφωνία που υπάρχει ήδη. Τονίσατε ότι υπάρχουν κάποια βήματα πρόοδου. Εμείς τα βρίσκουμε κάπως πιο οικονομικά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, από ότι εσείς. Γεγονός πάντως είναι ότι έχει σημασία το ότι υπάρχει ίδια η συμφωνία, διότι όπως λέχθηκε προηγουμένως, 60% των παγκόσμιων ενέργειων μεταφορών αφορά Ηνωμένε Πολιτείε και Ενωμένη Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι σε μια τέτοια εταιρική σχέση πρέπει να ισχύουν περίπου οι ίδιε ισότιμε δηλαδή συνθήκε. Δεν μπορεί κανεί να μιλήσει στην περίπτωση αυτή για κάτι τέτοιο όταν οι Αμερικανοί έχουν 49% μερίδιο στην αγορά μας και εμείς μόνο 25% στην δική τους. Είναι προφανής η έλλειψη ισορροπίας. Με μια μικρή αντιπροσωπή επισκεφθήκαμε την άνοιξη που μας πέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και προβήκαμε σε διαπραγματεύσεις και μας είπαν ότι αν θέλετε περισσότερη πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να επιτρέψετε για παράδειγμα νυχτερινές πτήσεις, θα πρέπει να κάνετε άλλες ρυθμίσεις για τον θόρυβο. Εμείς εξηγήσαμε ότι το θέμα εδώ σε εμά άπτεται της επικουρικότητας και ότι οφείλουμε να την σεβαστούμε. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε βέβαια άλλα πράγματα όταν θα έχουμε περίπου τις ίδιες ε, ρυθμίσεις. Μας είπαν λοιπόν τέσσερα πράγματα. Περιβάλλον, μπορούμε να πετύχουμε ορισμένα πράγματα και με το εμπόριο των εκπομπών. Ε, τα κοινωνικά πρότυπα έγιναν κάποια πράγματα, μιλήσατε και για δικαιώματα των επιβατών. Ανταγωνισμός, εκεί υπάρχει περιθώριο για πραγματική βελτίωση και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, έρχομαι ευθύ αμέσω στα δεδομένα. Οι Αμερικανοί έχουν διαφορετική αντίληψη περί προστασία προσωπικών δεδομένων και προσωπική σφαίρα από αυτήν που έχουμε εμεί. Εμεί βεβαίω θέλουμε να γίνει σεβαστή η προσωπική σφαίρα. Στην Αμερική είδαμε τα λεγόμενα body scanner. Είναι σύνηθε να έχουν εκεί αρχέ ασφαλεία όταν περνάει ο επιβάτη ολόκληρη η εικόνα του σώματό του. Ε, για μα εδώ πέρα αυτό είναι αδιανόητο. Θέλουμε οπωσδήποτε να προστατευτεί η προσωπική σφαίρα και τα προσωπικά δεδομένα και αυτά επίση πρέπει να γίνουν σεβαστά. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να τα συζητήσουμε και να τα μαζί σα και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχυμένο πλέον στι εξουσίε του από τη και τη Αγώνα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Δεν τήρησα τον χρόνο μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα όμως θα είμαι αυστηρός. Τον λόγο θα αναλάβει η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα... Μας χαροποιούσε όλους μια επιτυχής ε, συμφωνία και μετά από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων ε, έχει ήδη καθυστερήσει. Προφανώς αυτή η συμφωνία είναι μια πολύ σημαντική ε, πρόοδος και είναι ευπρόσδεκτη. Ε, με χαροποιεί το γεγονό ότι έγινε πρόοδο σε θέματα ασφάλεια και πρόσβαση αγορά, αλλά με απογοητεύει το γεγονό ότι δεν έχουμε ρυθμίσει πλήρω ε, τα θέματα τη ιδιοκτησία, του ελέγχου και του καμποτάζ. Επίση, είμαστε υπέρ ε, του κοινού ψηφίσματο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα θέματα εμπορία εκπομπών και με ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν ε, μπει στο κείμενο. Οι αεροπορικές ε, συμφωνίες έχουν ε, αναπτυχθεί μαζικώς ε, και είναι πολύ ευάλωτες στην Ευρώπη παρά την πρόοδο αυτή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα διαπραγματευτούμε χωρίς οποιοδήποτε τίμημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι δίκαιη, θα είναι στεναρή και θα οδηγεί σε πλήρη απελευθέρωση των αγορών που θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους αερομετοφερείς, τους καταναλωτές και τους Αμερικανούς φίλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Νάτρας. Α, δυστυχώς βλέπω ότι είναι απόν. Ερχόμαστε τώρα στο τμήμα της συζητήσεως που επιγράφεται Catch the Eye. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε και επίτροπε. Η Ένωση έχει ζητήσει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για αύξηση της ευελιξίας στην αγορά των αερομεταφορών με βάση και διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Η συμφωνία για τις εναέρειες μεταφορές ΕΕ, ΕΕ και ΕΕ, έχει καταλήξει σε μία προκαταρκτική φάση τον Μάρτιο και προβλέπει πλήρω άνοιγμα της αγοράς και δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία στις εναέριες μεταφορές και στη διαχείρισή τους ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ των αεροπλάνων και των προγραμμάτων μεταφοράς και να μειωθεί η αρνητική επίπτωσή τους στο περιβάλλον. Η μεταβιβάση των προσωπικών στοιχείων των επιβατών προς τις Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να βασίζονται και στη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και σε διεθνείς συμφωνίες που να έχουν νομοθετική ισχύ και να μην διαφέρουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Λυπούμαστε διότι οι ανταλλαγές των εκπομπών διοξιδίου δεν είναι τμήμα της προκαταρκτικής συμφωνίας και θα θέλαμε να γίνουν και άλλες διαπραγματεύσεις και για το θέμα αυτό μέχρι το 2012. Ορίστε για να καταλήξετε κύριε Χάτρα που ήρθατε. Όχι. Η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και ομιλήτριες για τα σχόλιά τους παρά την προκεχωρημένη ώρα βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ. Europe and United States together represent close to 60% of Γενικά οι ενέργειες μεταφορές είναι πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομίας και άρα και η συμφωνία αυτή όχι μόνο για τους πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ειδικότερα για τους επιβάτες και επιβάτριες. Εκτός από την αξία αυτή που είναι προφανής υπάρχει και το θέμα της σημασίας των ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο υπήρων γιατί είναι στρατηγικός εταίρος μας στις εναέρες μεταφορές ε, είπα. και θα έπρεπε αυτή η στρατηγική εταιρική διατελαντική σχέση να ενδυναμωθεί μετά από την πρώτη φάση για να υπάρξει η εγγύηση ενός σταθερού πλαισίου και των μελλοντικών σχέσεων. Αρκετοί ομιλητές και ομιλήτριες τόνισαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για να γίνουν κι άλλες και πρόσθετες πρόοδοι και πράγματι μία από τις επιτυχίες της πρώτης φάσης είναι ότι ακριβώς προβλέπει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να απαντήσω τώρα σε κάτι που είπε κάποιος συνάδελφος ότι φυσικά η Κομισιόν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνδικητής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο γιατί θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή του. Πολύ. Όταν υπάρξουν, δοθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η συμφωνία αυτή θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε από την κρίση. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Η Κομισιόν, όπως και πολλοί από τους ομιλητές και ομιλήτρες, συμφωνεί ότι η δεύτερη φάση της συμφωνίας δεν είναι τέλεια. Είναι πολύ σημαντική πρόοδος, αλλά δεν είναι τέλεια ή τελειωτική η, συμφωνία, η φάση αυτή της συμφωνίας. Θα θέλαμε κι εμείς να είχε αλλάξει ο Αμερικανικός νόμος για την ιδιοκτησία και διακυβέρνηση των Αμερικανικών αεροπορικών εταιριών αλλά δεν εξαρτάται αυτό από τις Αμερικανικές αρχές με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Μπορεί να την κάνει την αλλαγή αυτή μόνο το Κογκρέσο. Και εδώ έρχομαι να σας δώσω ένα σημαντικό μήνυμα. Η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη της την επιρροή για να πείσει και το Κογκρέσο για την ανάγκη αγκαιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και εδώ το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο με τις ευκαιρίες που έχει επαφών με τους Αμερικανούς βουλευτάς του Κογκρέσου δηλαδή. Ελπίζω να παίξετε το ρόλο αυτόν για να προχωρήσει ο διάλογος, οι συζητήσεις και ιδιαίτερα τα νομοθετικά βήματα που χρειάζονται. Για το θέμα που έθιξαν μερικοί ομιλητές τώρα, δηλαδή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα ήθελα να σας αναφέρω πληροφοριακώς ότι αυτό δεν αποτελεί τμήμα της Συμφωνίας των Εναερίων Μεταφορών, είναι θέμα εσωτερικό και δικαιοσύνης. Και φυσικά έχει τη σημασία του και θα ληφθεί υπόψη σοβαρά στις μελλοντικέ συζητήσεις. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Πρόεδρε να σταματήσω εδώ με την άδειά σας και σας ευχαριστώ εκ νέου για την επικοδομητικότητα αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία μου για την σύνοψη που κάνατε τη συζητήσεως. Έχουμε